αυτές ε, να συνεισφέρουν, πρέπει σίγουρα να αποφανθούμε ξεκάθαρα για την κατάσταση των κοπτών ε, χριστιανών. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι αυτό το οποίο ζητούσε το ΕΛΚ ήταν η ψηφοφορία να γίνει στη δεύτερη σύνοδο της του Οκτωβρίου, έτσι, σε δύο εβδομάδε. Αυτό έχω εγώ μπροστά μου. Ποιο θέλει να μιλήσει υπέρ αυτή τη πρόταση. Κύριε Σβόμποτα, ναι, εξαρτάται από το τι συζητάμε. Το γεγονό όμω είναι, κύριε Πρόεδρε,